αν δεν έχετε κάρτα δεν ψηφίζετε. Το έχω πει και στο παρελθόν. Επειδή είναι πολύπλοκη η διαδικασία χωρίς κάρτες, αποφασίσαμε ότι δεν θα δεχόμαστε τις ψήφους που δεν γίνονται με κάρτα. Λοιπόν, έχετε ελπίζω όλες τις κάρτες σας και όποιος δεν έχει να πάει γρήγορα να τη φέρει. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ε, προφορική ερώτηση της κυρίας Ζολή. Δεν υπάρχει τορκολογία, Μα κύριε Ντέβα, Σας το είπα κύριε Ντέβα, είχαμε πάρει απόφαση την προηγούμενη φορά. Δεν υπαναχωρώ. Δεν πρόκειται να ψηφίσετε σηκώντα το χέρι. Πολλές πολιτικές ομάδες συμφώνησαν, πήραμε την απόφαση αυτή, είπαμε ότι ήταν η τελευταία φορά τουλάχιστον 10 φορές έχει γίνει αυτό και την τελευταία φορά σας το είπα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να είμαι τόσο αυστηρή, αλλά το αποφασίσαμε. Όποιος δεν έχει κάρτα ψηφοφορίας δεν ψηφίζει. Το είπαμε, το αποφασίσαμε και ομόφωνα. Λυπάμαι, παραλυπάμαι, αλλά αλλιώς ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε έναν από τους βοηθούς σας για να σας φέρει την κάρτα σας. Το λέμε, το ξαναλέμε, είναι η δεύτερη χρονιά και πάλι δεν υπάρχουν κάρτες. Λοιπόν, κάποια στιγμή τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Προφορική ερώτηση της κυρίας Ζολή. Προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο χωρίς τροπολογίες. Ψήφι υπέρ. Α, ναι, βέβαια, ηλεκτρονικά, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. ομόφωνα δεκτή. Δεύτερη προφορική ερώτηση, χωρίς τροπολογίες, πάντα από την κυρία Ζολή, ηλεκτρονική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας ομόφωνα και πάλι δεκτή. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος ε, της κ. Ζολή, τροπολογία 3, διανατάσσος χειρός αυτή τη φορά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, παράγραφος 2, ε, σε, 4, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 2α, ε, 6, τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά θα το ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 9 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ συγκρίνει. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9 προς 9. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, δεν ξέρω. Να ελέγξουμε. Τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελογικές αναφορές, ε, citations, ε, στην 4, τροπολογία 1 και 2, ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνονται. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος υπέρ, κατά, ηλεκτρονικά, με συγχωρείτε, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας. Ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα. Περνάμε στον προϋπολογισμό χρηματοοικονομική υποστήριξη Αφγανιστάν. Κύριε Γκέρες, έκθεση, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απο... εγκρίνεται. Συγγνώμη λέει πρόεδρος. Τέταρτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 3. Υπέρ. Δεν είναι έτσι. Όχι, καλά τα λέω. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Την προφορική τροπολογία, ναι, την ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, Καταπίπτει αυτή. Λοιπόν, τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Όχι. Καταπίπτει. Καταπίπτει. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές δεν ξέρω. Ηλεκτρονικά. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά απόχέ. δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα επί του συνόλου, τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβολή της Επιτροπής ΔΕΒΕ Μπλα μπλα μπλα μπλα λέει πρόεδρος. Donc c'est pour Paris Jolie aussi. Comment Tu as la version française là. Ok. Alors. Lipon. Λοιπόν, παράγραφος 1, τροπολογία 8 στη ψηφορία για το πρώτο μέρος. Ε, ε, εγκρίνεται. Δεύτερο, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά να επαληθεύσουμε ηλεκτρονική ψηφορία για το δεύτερο τμήμα. Αρχή ψηφορίας, πέρα ψηφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, σε δύο τμήματα και πάλι. Σε τρία, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο για το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο μέρος, τι είπατε? Για το δεύτερο μέρος, ηλεκτρονική ψηφορία, ανέρξη. Ωραία, εγκρίνεται. Να σηκώνετε τα χέρια σας, κοιτάξτε, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τα ίδια συνεχώ Τρίτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Και δεν ξέρω. Ηλεκτρονική έναρξη. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. Δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 11 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι. Λοιπόν, για την 11 δεύτερο τμήμα ηλεκτρονική ψηφορία έναρξη. Πέρας ψηφορίας απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 14 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική έναρξη για την 14 πέρας ψηφορίας απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται, επαλήθευση ηλεκτρονική, έναρξη ψηφορίας για το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ για το πρώτο, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ κατά επαλήθευση ηλεκτρονική έναρξη ψηφοφορίας. Παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 20 εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική ψηφορία έναρξη πέρας ψηφορίας εγκρίνεται 22 υπέρ κατά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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα, ενέργηση πέρας, απορρίπτεται. Το για 4, υπέρ, κατά, αποχές επαλήθευση, ενέργεια ψηφορίας, για την τρία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. 4 με συγχωρείτε. τέσσερα υπέρ κατά αποχέ, Επαλήθευση και πάλι νομίζω ότι έχουμε μία ψήφο διαφορά. Ψηφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Επαλήθευση ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Όχι, μισό λεπτό. Ψηφίζουμε επί του συνόλου. Ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. 21 ψηφί υπέρ, 2 κατά. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία.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 La situation... Η κατηγορία, η κατάσταση. Α, κύριε Μπέμεν, ακόμη δεν ξεμούδιασε ο κύριος Μπέμεν. La situation des femmes en de... Η κατάσταση των γυναικών σε περίοδους πολέμου. είναι η κυρία Γκρέζ, Να δούμε τι γίνεται και με την Επιτροπή Γυναικών. Το αντικείμενο βεβαίω είναι η προστασία των γυναικών κατά κάθε μορφή βία, σεξουαλική και άλλη βία σε περίοδου πολέμου και η συμμετοχή από την άλλη μεριά των γυναικών σε όλε τι δραστηριότητε για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανασυγκρότηση των χωρών μετά από του πολέμου. Το αντικείμενο είναι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις γυναίκες και διαμόρφωση ανάλογα της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη. κυρία Γκρέζ θα παρουσιάσει το κείμενο. Ε, έχει περίπου 10 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, με την ε, γνωμοδότηση αυτή για τις γυναίκες σε περίοδους πολέμου προσπαθώ να πω το εξής. Καταρχήν το κείμενο συγγράφεται στον απόϊχο συναφών κειμένων και μας ενδιαφέρει πολύ διότι συνεχίζει να στέλνει το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε από την αρχή αυτής της εντολής. Δηλαδή, την ανάγκη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιτροπών. Η κατάσταση των γυναικών σε περίοδου πολέμου δεν αφορά φυσικά μόνο την Επιτροπή Γυναικών, αλλά και εμά. Εννοείται. Πιστεύω ότι η σεξουαλική βία είναι ανησυχητικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια περίοδων συγκρούσεων αλλά και μετά και γι' αυτό το λόγο ακριβώς θεωρούμε υποχρεωσή μας να μιλήσουμε για την κατάσταση των γυναικών αυτών κυρίως ε, από την σκοπιά της πρόληψης των συγκρούσεων. Στο κείμενο που έχετε μπροστά σας, με συγχωρείτε είμαι λίγο αδιάθετη και με την ισχύ σας κυρία Γκρέζ. Λοιπόν, το κείμενο που έχετε μπροστά σα. περιλαμβάνει αριθμό προτάσεων, συστάσεων που μόλις υπογραμμίσατε με σκοπό την ενίσχυση της συνειδητοποίησης της θέσης των γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη είχε αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις στον τομέα αυτών θα μπορούσα να υπενθυμίσω εν παρόδο την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 2011-2015 που συνοδεύει το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών επί του ίδιου θέματος. Παρά τις πρωτοβουλίες όμως αυτές, η πρόκληση αντιμετωπίζεται την πλευρά μας με τρόπο κατακαιρματισμένο. Η πρόκληση λοιπόν είναι να καταστρώσουμε μια πιο συνεκτική πολιτική στο πλαίσιο μεταξύ άλλων της εξωτερικής βοήθειας. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή μεταξύ της εξωτερικής ε, δράσης και της διαχείρισης κρίσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι Στόχο είναι προφανής, να εξασφαλίσουμε μεταξύ άλλων και πόρους για να ενισχύσουμε τις δράσεις μας υπέρ τη ισότητας και δι στον τομέα των χρηματοδοτικών μηχανισμών για την ανάπτυξη. Στις εκθέσεις που έχουμε στην διάθεσή μας διαπιστώνουμε ότι η στάση μας, η πολιτική μας τον της ανάπτυξης, η πολιτική μας για την ανάπτυξη δεν ενσωματώνει, δεν συμπεριλαμβάνει την πτυχή, την διάσταση γυναίκες. Στο κείμενο διαπιστώνεται επίσης ότι η πρότασή μας είναι να βελτιώσουμε τους σχετικούς δείκτες και να αξιολογούμε την κατάσταση όχι μόνο από ποσοτικής αλλά και από ποιοτικής απόψεως. Το θέμα είναι εξαιρετικά λεπτό. Οι αριθμοί δεν αρκούν για να περιγράψουν την κατάσταση. Χρειαζόμαστε και μια ποιοτική προσέγγιση. Μιλάμε για ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε. Και τέλος, εν κατακλείδη πριν να δώσω τον λόγο στους συναδέλφους, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε τη σημασία των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των αντιπροσωπιών ώστε να ευαισθητοποιηθούν για τα θέματα που έχουν σχέση με τα δύο φύλλα. Κατά τα υπόλοιπα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσ, Ο λόγος στην κυρία Κρατσίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια την κυρία Γκρές ε, για την πολύ καλή κατάσταση, την πολύ καλή έκθεση που ε, συνέταξε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το όσο έχει κάνει μέχρι τώρα, θα θέλαμε όμως ε, να προσθέσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ε, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία ε, στην πολιτική της ε, χώρας σχετικά με την περίληψη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές. Θεωρούμε ότι οι εκπρόσωποι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση των γυναικών σε, ε, περιοχές, ε, σε εμπόλεμες περιοχές. Αυτό ισχύει για την περίοδο 14 έως 2020. Ίσως μπορούμε να αναφερθούμε και στις ιδιαίτερες διατάξεις που προβλέπουν επιπρόσθετη προστασία των γυναικών από διασμό, από κάθε μορφή επίθεση, κυρίως όσον αφορά τις μητέρες και τις μητέρες νέων παιδιών, όσον αφορά τα τρόφιμα, ε, τα, την ενδυμασία, την ιατρική περίθαλψη, έτσι ώστε να αποφευθούν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και μεταδιδόμενες σεξουαλικές ασθένειες. Αυτά πάντα για την περίοδο 2013 έως 2020. Επίσης, Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι καταδικάζουμε ε, απερίφραστα την ε, ομοιρία κυρίως ε, γυναικών που βρίσκονται σε περιοχές, σε εμπόλεμες περιοχές. Απευθυνθήκαμε, κάναμε μια έκκληση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερες ε, τιμωρίες εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Ε, αυτό ισχύει για την Κεντριακή Αφρική, για το Σουδάν, για τον Νταρφούρ, για πολλές περιοχές. Πρέπει να υπάρχει καλύτερος ε, συντονισμός με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι οι συγγενείς έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν πληροφορίες για τους αγνοούμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα παρέμβω ίσως αργότερα και πάλι. Ο κύριος Μαρτίνεθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι άκρος ενδιαφέρουσα η έκθεση. Πρώτα απ' όλα το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι και δραματικό και άκρος επίκαιρο. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ σωστή και την προσέγγιση της κυρίας Γκρέζ. Είναι σαφές ότι η Επιτροπή μας έχει ρόλο και λόγο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα ήταν επικίνδυνο να θεωρήσουμε ότι το ζήτημα αυτό αφορά την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής για την Ισότητα, για τα δικαιώματα των γυναικών. Νομίζω ότι εμπίπτει και στο δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων και φαντάζομαι και κάποιες άλλες επιτροπές μπορούν να γνωμοδοτήσουν για το ζήτημα αυτό. Όλοι γνωρίζουν ότι οι γυναίκες σε τέτοιες ε, καταστάσεις είναι πολύ περισσότερο θύματα από οποιονδήποτε άλλον. Είναι θύματα πολέμου Σίγουρα, όπως οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, οι άνδρες, ε, οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο όν ζει υπό τέτοιες συνθήκες, αλλά όπως καταγγέλλεται και είναι γνωστό, οι γυναίκες είναι θύματα ακριβώς επειδή είναι γυναίκες, λόγω του φίλου τους. Ως γυναίκες, ως μητέρες, ως άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους και παιδιά. Είναι θύματα δηλαδή ακριβώς επειδή ασχολούνται επειδή φροντίζουν άλλους τομείς της κοινωνίας, που και αυτοί είναι θύματα του πολέμου. Επίσης βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι οι σεξουαλικές κακοποίησεις γίνονται ένα εργαλείο ε, πολεμικό, ένα όπλο και αμοιβή των ιστοφόρων. Και δεν είναι μόνο η Αφρική. Έχουμε δει πριν κάνα δύο-τρεις δεκαετίες πολέμους και επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η κατάσταση των γυναικών ήταν η ίδια με την κατάσταση των γυναικών στην Αφρική και εκεί ήταν θύματα και μεταξύ άλλων σεξουαλικής κακοποίησης συστηματικής. Τις χρησιμοποιούσαν ως όπλο πολέμου για τα τακτικά στρατεύματα αλλά και για τα άτακτα εντό αγωγικών στρατεύματα τις περισσότερε φορές. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Γκρέσ και να της πω ότι και θα στηρίξουμε την έκθεσή της και θα συνεργαστούμε μαζί της. Πιστεύω ότι λείπει κάτι και καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Και συγκεκριμένα μιλώ για τη σημασία που έχει να συνεργαστούμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στενά με τα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη στον τομέα αυτό πραγματικά έχουν σημαντικό έργο. Η δράση τους είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα έχει στεφθεί και με αρκετή επιτυχία σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Έχω και οικογενειακή σχέση ε, με κάποιο άτομο που εργάζεται στον τομέα αυτό. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι επικεντρώνονται βέβαια τελευταία στην Αφρική, στον ΟΗΕ, αλλά έχουν ασχοληθεί και με άλλες χώρες όπως ήταν η Καμπότζη πρόσφατα. Νομίζω ότι πρέπει και να στηρίξουμε αλλά και να βασιστούμε σε αυτό που κάνουν ε, τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό θα είχε πολύ ευεργετική ε, επίπτωση ε, και για τη σημασία της έκθεσης που θα εκπονήσει η κυρία Γκρέσ και την οποία ελπίζω να εγκρίνουμε με μια μεγάλη πλειοψηφία ή καλύτερα ακόμη και με ομοφωνία. Ευχαριστώ και ακόμη μια φράση χαρητήρια στην κυρία Γκρέζ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Μαρτίνεθ. Η κυρία Σνίμπερ Γέστραμ τώρα έχει το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ ε, για αυτή την τόσο σημαντική έκθεση που κατά την άποψή μου όπως έχει ληφθεί και από τους υπόλοιπους είναι πάρα πολύ καλή. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καταρχήν στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, στην ε, υποστήριξη που ε, παρέχεται σε τοπικές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό θα πρέπει να διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, κυρίως για τις ομάδες γυναικών, ε, που έχουν μια πολύ συγκεκριμένη μερίσια διάταξη. Δηλαδή η βελτίωση του ε, προς εκμετάλλευση παρεχόμενου δυναμικού είναι πολύ σημαντικό. Κυρίως ε, στις εμπόλεμες περιοχές γιατί δεν υπάρχει κατ' ουσίαν η παρουσία του κράτους. Έτσι λοιπόν οι οργανώσεις γυναικών μπορούν αν έχουν αυτή τη βοήθεια να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε αναπτυξιακά προγράμματα από γυναίκες για γυναίκες διότι οι ίδιες οι γυναίκες ε, δεν είναι μόνο το αδύναμο φύλλο, οι γυναίκες ε, είναι και πάρα πολύ δυνατές. Ένα δεύτερο θέμα είναι η πρόσβαση των γυναικών ε, σε ιδιοκτησία γης. Μετά από σειράξεις οι γυναίκες, κυρίως οι διαζευγμένες και οι χείρες, πολλές φορές έχουν πρόβλημα να γυρίσουν στην πατρίδα τους και να αποκτήσουν και πάλι γη. Ε, λόγω του ρόλου των γυναικών σε ορισμένες κοινωνίες, αυτό είναι το ένα, και κατά δεύτερον λόγω του ότι στις χώρες αυτές και μετά το πέρας των σειράξεων εξακολουθούν να υπάρχουν εχθροπραξίες. Ε, ε, καταστρέφεται ο πολιτισμικός ιστός, αλλά παρόλα αυτά μπορεί κανείς να βοηθήσει μια κοινωνία η οποία κοινωνία ε, δίνει πλέον τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν ε, γη στην διοκτησία τους και γενικότερα να συμμετέχουν στην κοινωνία. Εδώ λοιπόν σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς να βοηθήσουμε τους φορείς αυτούς. Και κάτι άλλο πρέπει να έχουμε κατά νου. Την παροχή βοήθεια σε πρωτοβουλίες ε, που μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες γυναικείων, γυναικών υποψηφίων. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τους άντρες, άρα δηλαδή πρέπει να κινητοποιήσουμε και τους άντρες σε όλα τα επίπεδα. Οι άντρες οφείλουν να κατανοήσουν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών θα συνεπάγεται και για αυτούς ε, μεγάλο κέρδος. Νομίζω σήμερα το βράδυ ε, λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες που σημαίνει ότι θα έχουμε ακόμα κάποιο χρόνο να καταθέσουμε ίσως ορισμένες. Η κυρία Θεοχάρους παρακαλώ. Είναι όντως πολύ σημαντική η αναφορά που έχει παρουσιαστεί σήμερα. Ε, και θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την ε, ραπορτέρ. Ε, θα συμφωνήσω όμως ότι κάτι λείπει και αυτό είναι οι πραγματικές συνθήκες του πολέμου και οι εμπειρίες που βιώνουν οι γυναίκες αυτές ε, αν ειδωθούν μέσα από τον ρόλο της Επιτροπής Ανάπτυξης στη διαδικασία του εκδημοκρατισμού των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, των αναπτυσσομένων χωρών, στη διαδικασία ανάπτυξης δημοκρατικής παιδείας και κουλτούρας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι ένας μηχανισμός τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως Επιτροπή. Τώρα, το τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, από τη στιγμή που θα εκραγεί ένας πόλεμος, είναι όντως ε, μια βάρβαρη καταπίεση των δικαιωμάτων των γυναικών, γιατί η γυναίκα έχει την ευθύνη της προστασίας των παιδιών κυρίως και των γερόντων, αλλά και υφίσταται όλα τα προβλήματα που υφίσταται ο γενικός πληθυσμό. Για παράδειγμα, δεν σταματούν οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν επειδή κάποιοι πολεμούν στην πρώτη γραμμή. Όταν ε, υπάρχει ήδη ένας διαχωρισμός, πρέπει να έχουν όλες οι γυναίκες πρόσβαση στους μηχανισμούς βοήθειας. Δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Οι γυναίκες οι οποίες καλούνται οι ίδιες να πάρουν τα όπλα και να πολεμήσουν, δεν συνάδει με την δεν θα ήθελα ότι να πω ότι συνάδει με την ανδρική φύση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συνάδει ιδιαίτερα με την γυναικεία φύση να παίρνει τα όπλα η γυναίκα και να ε, στέλνεται στην πρώτη γραμμή. Ε, δεν έχει την εκπαίδευση για να προστατεύει τον εαυτό της, τα παιδιά της, αυτούς που φροντίζει κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής ε, επιχείρησης. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το εντάξουμε μέσα στο ε, στο report και παράλληλα να δούμε αν πρέπει να κληθούν κάποιες χώρες να υπογράψουν τη συνθήκη της Ρώμης του 1998 όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για την προστασία των γενικών από σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια των πολέμων καθώς επίσης και για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Ινστιτούτου το οποίο θα παρέχει ψυχολογική, νομική, ε, βοήθεια στις γυναίκες οι οποίες είναι θύματα σεξουαλικής ή άλλης βίας κατά τη διάρκεια των πολέμων. Αυτά σαν αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Κάσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφός μου από δεξιά προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή της ε, γραμματέως ή της γραμματίστας που αν φαίνεται το κατάφερε. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι ένας από τους άνδρες της Επιτροπής, ε, θέλω ε, να εκφράσω τις ανησυχίες μου σε αυτές που ήδη εκφράστηκαν για τα θέματα των γυναικών. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Βλέπουμε να υπάρχει όλο και περισσότερο το θέμα του εκδικητικού βιασμού ε, και στις ε, λεσβίες πριν, ε, κατά και μετά τις σειράξεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε επιγόντως αυτό το θέμα. Κυρίως στα ψηφίσματα που θεσπίζονται μετά την επίτευξη ειρήνης οι γυναίκες ε, καλούνται να ανοικοδομήσουν τις οικογένειες ε, και ε, τις πατρίδες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό είναι κάτι που το ανέφερε και ο κ. Μπέρμαν. Δηλαδή, χρειαζόμαστε έναν ύπατο εκπρόσωπο που να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Γιατί εγώ το βρίσκω πάρα πολύ περίεργο ε, το γεγονός ότι στην Επιτροπή μας ε, δεν έχουμε κανένα που να εκπροσωπεί αποκλειστικά και μόνο ε, το θέμα της ισότητας ε, των δύο φύλων και της ταυτότητας των δύο φύλων. Ίσως να κάνω λάθος, αλλά κατά την άποψή μου εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τόσο επίγον και σημαντικό θέμα και συνεχίζουμε να μιλάμε για τη διάσταση του φύλου και την κατάργηση διακρίσεων. Αλλά πού είναι άραγε ο άνθρωπος αυτός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι αρμόδιος για όλα αυτά. Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι απλά επανανακαλύπτουμε τον τροχό. Δηλαδή επαναρχόμεθα στα ίδια και τα ίδια ψηφίσματα Βασικά όμως ξεχνάμε ότι μιλάμε εδώ για θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα λοιπόν ερώτημα που θέτω είναι γιατί όλα αυτά αγνοούνται από το Σώμα των Επιτρόπων. Ούτε ένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Και θέλω επίσης να πω, ε, κυρία Άστον, παραδείγματο χάρη, δεν χρειάζονται χρήματα. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί ε, πρώην διπλωμάτες, ας μείνουν εκτός οι πολιτικοί, οι οποίοι μπορούν στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης να αναλάβουν το θέμα αυτό, να ορίσουν έναν ύπατο εκπρόσωπο για την ισότητα των δύο φίλων και την κατάργηση των διακρίσεων. Ε, πρέπει να καταθέσουμε ένα αίτημα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και στην κυρία Άστον, ε, γιατί η ίδια λέει ότι δεν έχει τα απαραίτητα κονδύλια και ως εκ τούτου αυτό οδηγεί σε πάρα πολλά λάθη. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν τη δουλειά να τη μοιράσουμε σε όλους, να την αναλάβουν πολλοί. Επανέρχομαι όμως και πάλι σε αυτό που είπα στην αρχή. Όταν ήρθα για πρώτη φορά εδώ, πρέπει να σας πω, θεώρησα παντελώς απαράδεκτο το ότι ε, δεν υπάρχουν μόνιμοι εισηγητές. Εισηγητές ε, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, μια μικρή γραμματεία, που να ασχολείται μεταξύ άλλων με την ισότητα των δύο φύλων, ε, την κατάργηση των διακρίσεων με βάση το πρώην άρθρο 13, το, τώρα το νυν 19. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος να επιληφθεί αυτών των ε, θεμάτων, να προβάλλει τις αξίες μας, να φροντίζει για νομοθετήματα, για δράσεις, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, τότε ποτέ δεν θα γίνουμε μια επιτυχημένη οικονομική κοινότητα. Και τι θα γίνει αν αποτύχει και αυτό, απολύτως τίποτα. Δεν θα έχει απομείνει τίποτα. Εσείς τώρα κύριε Μπέρμα έχετε το λόγο. Πράγματι Πιστεύω ότι η κατάσταση των γυναικών ε, σε εμπόλεμε περιοχές είναι τόσο σοβαρή που άλλωστε θύματα και παιδιά, παιδιά και γυναίκες είναι στο μεγαλύτερο βαθμό ε, αυτών των καταστάσεων και είναι και στο στόχαστρο ε, για να εκφοβιστεί και να τρομοκρατηθεί ένας λαός. Ναι, ασχολείται η εθνική κοινότητα, αλλά νομίζω ότι σημαντικό και απαραίτητο θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει ειδικό εντεταλμένο εκπρόσωπο, όπως λέει ο Μάικλ, ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν τόσα χρηματοδοτικά μέσα και τόση πολιτική τομή, οι οποίοι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να δικαιολογείται ο ορισμός ενός ειδικού απεσταλμένου, ο οποίος θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό ή βασικό στόχο την ε, συνοχή των δράσεων, στόχο την προστασία των γυναικών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ένα υπόδειγμα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα έχει συζητηθεί σε όλες του, τις διαστάσεις και ήδη υπάρχει μια δεύτερη έκθεση από την Επιτροπή Γυναικών. Υπήρξε και κατά την προηγούμενη θητεία, είχαμε μια παρεμφερή έκθεση. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ ε, δυστυχώς δεν έχουμε γνωμοδότηση. Κατόπιν τούτου οι συνέπειες, ε, τα συμπεράσματα που εξάγαμε δεν είναι δεσμευτικά. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι έχουμε ε, εμπλακεί σε ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε ε, απαριθμίσει τα προβλήματα. Υπάρχει κάποια πρόοδος, υπάρχει κάποια βελτίωση και νομίζω ότι ε, τα επιχειρήματά μας ε, δυστυχώς ε, δεν πείθουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αν τελικά υπάρξει Οποτεδήποτε υπάρχει σύραξη, πάντα οι γυναίκες θα είναι θύματα. Το πρόβλημα θα παραμείνει άλυτο. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος, παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν τα Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς βλέπουμε τις γυναίκες να εξακολουθούν να υποφέρουν ως μητέρες. Τις βλέπουμε να είναι θύματα σεξουαλικής βίας και δυστυχώς και οι γυναίκες υποφέρουν προσπαθώντας να διεκπαιρεώσουν τον οικοκυριό τους. Μένουν μόνες τους με τα παιδιά τους πολλές φορές μετά τον πόλεμο γιατί πεθαίνουν οι άνδρες τους. Ε, μπορούμε να παριθμίσουμε λοιπόν πάρα πολλές τέτοιου καταστάσει. Ε, καταστάσεις. Ε, ίσως μπορούμε να καταρτήσουμε έναν κατάλογο και να αναφέρουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπουμε <clears throat> στη Βόρεια Αφρική, κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης, ότι πολλές γυναίκες αντιστάθηκαν και κατόπιν τούτου θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην ε, γυναίκα που κέρδισε ε, το βραβείο Νόμπελ στην Ιεμένη και αυτό μου άρεσε ιδιαίτερα το ότι δόθηκε το βραβείο Νόμπελ σε μια γυναίκα. Ευχαριστώ πολύ. Είστε ο λόγος στην Κομισιόν, κύριε Βαλπής. Το όνομά μου είναι Έλενα Βόλπη από την ΔΕΦΚΟ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή και κατ' ουσίαν ε, συμφωνούμε με όλα τα συμπεράσματα της έκθεσης. Ε, ήδη μας έχει προσφερθεί ευκαιρία να κάνουμε τα σχόλιά μας. Και κυρίως όσον αφορά τα σημεία εκείνα που υπογραμμίζουν το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των γυναικείων οργανώσεων, ε, των υποστηριχτών της ισότητας των δύο φύλων, πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις ε, για την ειρήνη και στην ε, κατοχήρωση της ειρήνης. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η σεξουαλική βία. Ε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα απλά να σας αναφέρω τι ακριβώς κάνουμε και εμείς για να συμβάλλουμε στην ενίσχυση δράσεων ε, σε αυτούς τους ε, τομείς. Όπως τα γνωρίζετε, το 2010 το Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των ε, δύο φύλων και αναφέρομαι σε αυτό το σχέδιο γιατί υπάρχουν αρκετοί στόχοι που έχουν άμεση σχέση με την κινητοποίηση ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων ε, με την βελτίωση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Ε, θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς ε, στην εφαρμογή του του 1325 των ΗΕ και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η βία που ασκείται εις των γυναικών. Πρέπει βεβαίως να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα εργαλείο, ένα μέσο αν θέλετε, ε, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα της τάξης του 1 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά όλες τις περιοχές, οι πολλές περιοχές καλύπτει Νότια Ασία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, ε, το Νότιο Κάφκασο, Γεωργία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και την Κεντρική Ασία, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν και Κυργιστάν. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό συνεχίζεται και κατ' ουσίαν είναι ο και ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να στηρίζονται οι ενέργειες ε, των γυναικείων οργανώσεων ε, και να εφαρμόζεται κυρίως ε, το ψήφισμα 1025 και άλλα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Κατόπιν, με το μέσο σταθερότητας υπάρχει και άλλο ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση τελικής διατύπωσης και πρόκειται κατ' ουσίαν για ένα πρόγραμμα, με συγχωρείτε, ξέχασα να εφαρπώ ότι το πρόγραμμα EDGR ε, εφαρμόζεται από νέες γυναίκες. Ένα άλλο πρόγραμμα που είναι σε φάση επεξεργασίας είναι μια γυναικεία πρωτοβουλία ε, με την, σε συνεργασία με την UNDP, τον Φορέα των Ηνωμένων Εθνών και πρόκειται πάλι για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί υπό το πρόγραμμα ε, δράσεις ε, του 2012 ε, υπό την αγίδα του Μεσίου Σταθερότητας και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ε, δυνατότητες των ΗΠΑ και την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 όπως επίσης να υπάρχει και πιο συντονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα δύο προγράμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κατόπιν ένας από τους ε, στόχους ε, του ε, προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δύο φύλλα, ένας από τους στόχους είναι να χρησιμοποιούμε ως το δυνατόν καλύτερα καλύτερα τα θεματικά μας προγράμματα, το εργαλείο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα θεματικά προγράμματα για να κινητοποιήσουμε τοπικούς πόρους έτσι ώστε αφενός ε, να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή του ψηφίσματος του 1325 αλλά και αφετέρου να μεριμνήσουμε για την εφαρμογή των δικών μας οδηγιών που έχουν ε, στόχο την ε, καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Σας παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να τελειώνετε σιγά σιγά γιατί έχετε ξεπεράσει το χρόνο που σας είχε, που είχε διατεθεί για σας. Τώρα λοιπόν είμαστε στην φάση της συγκέντρωσης των εκθέσεων και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν τοπικές πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο κυρίως όσον αφορά τα θεματικά προγράμματα. Ευχαριστώ πολύ και κρέας για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που υπενθύμησε τα άλλα τρέχοντα προγράμματα. Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν πλήρης, πολύ ενημερωτική. Άκουσα ότι παρά τα άλλα τρέχοντα προγράμματα πρέπει, όπως άλλωστε της το τόνισε, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσταση των γενικών σε περίοδους πολέμου. Σημείωσα και τα σημεία στα οποία πρέπει να βελτιώσουμε το κείμενο ιδιαίτερα το σημείο το οποίο αναφέρει η κυρία Κρετού όσον αφορά το θέμα των βιασμών και της πορνείας, καθώς και την ιατρική πτυχή του θέματος. Ο κ. Μαρτινές υπενθύμησε μάλιστα πως ο βιασμός γίνεται εργαλείο πολέμου σε εμπόλεμες περιόδους. Το αναφέρουμε και αυτό. Και άκουσα και άλλες συγκεκριμένες προτάσεις από τους συναδέλφους όσον αφορά για παράδειγμα τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη ή την ανάγκη υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Άκουσα επίση κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι πρέπει να δούμε τις γυναίκες όχι μόνο ως θύματα, για να τις προστατεύσουμε δηλαδή, αλλά και ως παράγοντες ανοικοδόμης μιας χώρας. Και αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Άκουσα επίσης μια άλλη πρόταση η οποία θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να ενσωματώσουμε στο κείμενο, είναι το δικαίωμα ιδιοκτησίας των γυναικών στην έγκυο ιδιοκτησία, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί σε πολλές περιοχές του κόσμου και πολύ ενδιαφέρον βεβαίω. Τέλος, η πρόταση του κυρίου Κάσμαν, και αυτή μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, να προσπαθήσουμε δηλαδή να ζητήσουμε, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό βεβαίω, αλλά να ζητήσουμε έναν, τη δημιουργία θέση ενός εκπροσώπου για τα θέματα αυτά. Τέλος, άκουσα και για το βραβείο Νόμπελ που πήγε σε γυναίκες της Ιμένης και της Λιβερίας. Είχαμε όντως εμπόλεμες καταστάσεις στις οποίες οι γυναίκες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο ενδεχομένω να προσκαλέσουμε αυτέ τι γυναίκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια στιγμή. Εν κατακλείδη, έχουμε προτάσεις, έχουμε ενδιαφέροντα σχόλια. Το ερώτημα το οποίο παραμένει είναι πώς οι αποφάσεις αυτές, οι προτάσεις αυτές θα γίνουν δεσμευτικές. Αυτό ακριβώς θα συνεχίσει να μας απασχολεί σας ευχαριστώ πολύ. Θα καταγράψουμε πολύ μεγάλη προσοχή περαιτέρω σχόλια ή ιδέες. Πολύ ωραία. Η προθεσμία λίγη σήμερα στις 5 για την υποβολή τροπολογιών. Οπότε, 7 Νοεμβρίου θα τα ξαναπούμε για την έκθεση. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει. αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης στο Νότιο Σουδάν. Παρουσία του ειδικού ανεταλμένου της ΕΕ για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν και μέλλον της ΑΦΕΤ. Ο Νικολό Ρινάλντι και ο κ. Στυρολία ήταν στο Νότιο Σουδάν 19 με 21 Ιουλίου του 2011 Στι 9 Ιουλίου, όπω ξέρετε, ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν, που ανεξαρτοποιήθηκε από το Σουδάν μετά από δεκαετίες εμπόλεμη κατάσταση με πολλά θύματα. Το κράτο αναγνωρίστηκε βεβαίω από τη διεθνή κοινότητα. Τα προβλήματα όμω παραμένουν. Η οριστική χάραξη των συνόρων μεταξύ Σουδάν και Νοτιού Σουδάν είναι αντικείμενο σειράξεων στην περιοχή και βέβαια δεν έχει λυθεί το θέμα του διαμοιρασμού των εσόδων από το πετρέλαιο. Η κυρία Μάρσεν είναι ειδική επιστελμένη της ΕΕ στο Σουδάν και τον Νότιο Σουδάν ε, και θα μιλήσει μετά από τον Πατριστή ο οποίος θα μας ε, πει λίγα λόγια για τις εντυπώσεις του από την περιοχή. Παρακαλώ να τηρήσετε τις προθεσμίες, το χρόνο μιλίας, γιατί έχουμε καθυστερήσει ο κ. Στυριλία για 8 λεπτά. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, το, Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε αποστολή μας στο Σουδάν τον περασμένο Ιούλιο. Είχα την τιμή να προεδρεύω της πολύ μικρής μας αντιπροσωπείας Μόνο ο κύριος Ρινάλντι με συνόδευσε κατά τη διάρκεια του δευτέρου μέρους της επισκεψής μας στην περιοχή. Δεν ήταν οι καλύτερες ε, συνθήκες και δεν μιλώ τόσο για τις συνθήκες ε, φιλοξενίας. Πάντως, είχαμε την ευκαιρία τουλάχιστον να διαπιστώσουμε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νέο κράτος. Στόχο τη αντιπροσωπεία μα ήταν να συλλέξουμε πληροφορίε για την ειρηνευτική διαδικασία, για τι ανάγκε τη διαδικασία ανάπτυξη, τη καλή διακυβέρνηση και να δούμε επιτόπου πω υλοποιείται η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν σα μιλήσω για τι παρατηρήσει μα, τι διαπιστώσει μα, θα ήθελα εκ μέρου τη μικρή μας αντιπροσωπεία να ευχαριστήσω κυρίως την κυρία Μάρσεν, την ειδική απεσταλμένη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, η οποία μα τιμά σήμερα με την παρουσία τη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το προσωπικό στη Τζούμπα για την πολύτιμη συμβολή του στην ε, ομαλή διεξαγωγή της αποστολής μας. Στις 9 Ιουλίου, όπως γνωρίζετε, η Δημοκρατία του Νοτιού Σουδάν έγινε το 189 ο ο μέλος των Ηνωμένων Εθνών και μέλος της ε, Αφρικανικής Ένωσης. Το μεγαλύτερο κράτος της Αφρικής είναι πλέον χωρισμένο σε δύο κράτη, μετά από δύσκολες περιόδους εμπολέμων σειράξεων, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανοικοδόμηση της περιοχής. Παρά το γεγονό ότι οι στατιστικές επιβεβαιώνουν ότι ο 35% για παράδειγμα των ενηλίκων είναι αναλφάβητοι, η πείνα είναι πρόβλημα, το οδικό δίκτυο έχει μόνο 50 χιλιόμετρα ασφαλιστωμένων δρόμων και τα δίκτυα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα. Δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης κλπ. Με σχεδόν ε, παντελή έλλειψη γιατρών, ε, μευτήρων, μεών κλπ. Το νότιο Σουδάν ζει ακόμη σε συνθήκες βίας, ε, συνθήκες εμπολεμού σύραξης. Νέα στρατητικά σώματα εμφανίζονται συνεχώς και οι σειράξει συνεχίζονται με εκατοντάδε νεκρούς. Το Νότιο Σουδάν Δυστυχώ φαίνεται ότι θα παραμείνει επί χρόνια υπό διεθνή εποπτεία και θα χρειάζεται βοήθεια από την πλευρά μα Το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων και αν συμπεριλάβουμε και την περίοδο από το 2003, η βοήθεια αυτή ανέρχεται σε πάνω από 760 εκατομμύρια. Τον περασμένο Μάιο εγκρίναμε επιπλέον βοήθεια 200 εκατομμύριων ευρώ για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια τριετούς περίοδου. Είχαμε πολλέ διμερείς συναντήσει στην περιοχή. συνέντηση με την κυρία Μάστεν, η οποία θα έρθει, φαντάζομαι, αργότερα θα μας μιλήσει για την αποστολή της. Μιλήσαμε με την μικρή νέα εθνοσυνέλευση, με τον υπεύθυνο γραμματέα για την ειρηνευτική διαδικασία, με τον Επίτροπο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, στους εκπροσώπους του ΟΗΕ, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από την περιοχή. Και Άστεν συζήτησε δύο θέματα κυρίως, τον ρόλο της Κίνας στην περιοχή και το θέμα της ασφάλειας. Όσον αφορά την Κίνα, δεν θα είναι έκπληξη να σας πω ότι έχουν έρθει οι Κινέζοι με πολύ μεγάλη όρεξη στην περιοχή για πετρέλαιο και για τον ορεικτό πλούτο της περιοχής. Επ' αυτού, κύριε Μάστερ, ε, σε σύνεση και μια συνεργατική προσέγγιση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινέ ε, θέσεις ως προς το θέμα. Εκφράσαμε την ανησυχία μας όσον αφορά την, τα δικαιώματα του ανθρώπου και το περιβάλλον που δεν γίνονται αντικείμενα φυσικά ιδιαίτερου σεβασμού στο πλαίσιο τη συμφωνία με την Κίνα. Στην ασφάλεια, στον τομέα τη ασφάλεια, διαπιστώσαμε ότι γίνεται σημαντική προσπάθεια για την βελτίωση τη κατάσταση, κάτι το οποίο είναι προπόθεση για την ειρήνη και την βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτό υπογράμμισαν και άλλε προσωπικότητε στην περιοχή. Η κυρία Μάρστεν ε, υπογράμμισε ότι η αποστατιωτικοποίηση είναι βασική προπόθεση στην περιοχή για τη νέα κυβέρνηση αφιερώνει ένα μεγάλο μέρο του προπολογισμού στι θεωρητικέ δαπάνε. Ο στρατό είναι 140.000 άνθρωποι. Η επανένταξη του πληθυσμού στην ε, κοινωνία είναι ένα θέμα, όπω και θέμα είναι η απασχόληση και, και δι τη απασχόληση των ε, πρώην στρατιωτών στο πλαίσιο της νέας κοινωνίας των πολιτών. Μιλώντας με άλλους εκπροσώπους θεσμών της περιοχής, διαπιστώσαμε ε, ότι πολλά θέματα εκκρεμούν όπως ο, ρόλος του Σουδανικού Κοινοβουλίου στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης δημοκρατίας. Το Γραφείο για την Πραγωγή της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας που συνόδευε την αντιπροσωπεία υπενθύμησε όλες τις ευκαιρίες συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας στην περιοχή. Οι ερευνητικές συνομιλίες συζητήθηκαν επίσης. Υφίστανται πολλά εμπόδια, εννοείται. Μεταξύ αυτών η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, ορισμός των συνόρων. Το θέμα της διαχείρισης των πόρων και δι του πετρελαίου. Όσον αφορά την προβληματική της ασφάλειας, πέρα από το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη. Διάφοροι πόλεμα στην περιοχή συνεχίζουν σε κινητοποίηση. Σημειώνονται συνεχώ διάφορε εξηγέρσει που καθιστούν την κατάσταση εύθραυστη. Τα Ηνωμένα Έθνη υποστηρίζουν μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, την δημιουργία ενό ε, κρατικού ταμείου στο οποίο η κυβέρνηση θα επενδύσει ένα μεγάλο μέρο των εσόδων του πετρελαίου. Το ταμείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένε επενδύσει. Η χάραξη των συνόρων βεβαίω συζητήθηκε και αυτή κατά επανάληψη γιατί η χάραξη των συνόρων θα επηρεάσει το θέμα τη μετακίνηση των πληθυσμών καθώ και το θέμα τη κατανομή των πόρων προ το πετρέλαιο. Όσον αφορά την ε, ορθή διακυβέρνηση και το κράτο δικαίου, ακούσαμε προσεκτικά τον εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο οποίο ε, μα είπε ότι δεν είχαν γίνει αρκετά τον τελευταίο χρόνο υπέρ της κοινωνίας των πολιτών. Μας είπε επίση ότι υπάρχει η έλλειψη ενημέρωσης της, ε, από την κυβέρνηση. Τα θέματα όλα αυτά είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Από την άποψη της ασφάλειας η κατάσταση είναι εκρηκτική. Η φτώχεια είναι απίστευτη και να ζητούμε μια οριστική λύση για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν την κατάρτιση, την κατάστρωση ενός εθνικού σχεδίου που προβλέπει θεσμούς για να μπορέσει η χώρα να αναπτυχθεί. Επιπλέον το πετρέλαιο και τα ορυκτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο αντί για πλεονέκτημα, γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομέ ούτε το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε το πρόβλημα αυτό της διακυβέρνησης, το θέμα της διαφθοράς, να μην αναστείλουν την ανάπτυξη, να μην αποτελέσουν εμπόδιο για το νέο κράτος, να μπορέσει να επιβιώσει το νέο κράτος ως μέλος της διεθνούς κοινότητα. Επ' αυτού από τις επαφέ μας με τους ε, επισήμους με την σημασία του διαλόγου και της συνεργασίας την ένταξη του νέου κράτους στη Συμφωνία Κοτονού η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδαματίσει το σημαντικό ρόλο και το ίδιο ισχύει και η διεθνής, η διεθνή ε, κοινότητα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τριλή, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγο στην κυρία Μάτσεν για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ιδιαίτερα επικοδομητική ε, εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνάντησα στην Τζουμπάντ. Ε, στην Τζούμπα, στην πρωτεύουσα, στις 9 Ιουλίου είχαμε την ανεξαρτησία της χώρας, τις ε, εορτές για την ανεξαρτησία της χώρας, για την ανεξαρτησία που απέτυχε με πολύ μεγάλο κόπο η χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να βοηθήσει σε αυτήν την ανεξαρτησία, έτσι ώστε το σύστατο κράτος να αποκτήσει την ευημερία του και να μπορεί να ανταποκριθεί ε, στις προσδοκίες ε, των πολιτών. Εξέφρασε λοιπόν η, η εκπρόσωπος τις ευχές της και έφτιασε θεμέλια έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρεις μήνες μετά την ανεξαρτησία ο πρόεδρος Κύρ, Κύρ ε, ε, συνέστησε το Υπουργικό του Συμβούλιο. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά την ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά εξακολουθεί η κυβέρνηση να έχει αντιμετωπίσει πολλά και δύσκολα καθήκοντα, κυρίω όσον αφορά το πρόβλημα τη ε, υπανάπτυξη ε, και το γεγονό ότι δεν υπάρχουν αρκετέ δυνατότητε για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα όπω είναι η βία ανάμεσα στι ε, φυλέ, δεν μπορούν να απορροφηθούν όλε αυτέ οι χιλιάδε ανθρώπου που επιστρέφουν από το βορρά. Επίση, ψηλέ τιμέ τροφίμων, πληθωρισμό μετά την εισαγωγή του νέου νομίσματο και τον εμπορικό που επιβλήθηκε στα σύνορα. Υπάρχουν και ανθρωπιστικές προκλήσεις που έχουν σχέση με την επισητιστική ασφάλεια και με την εισρωή των εκτοπλισμένων από τις σειράξεις που υπάρχουν στην περιοχή. Εξάλλου, εξακολουθεί να υπάρχει ένταση με το Βορρά, γιατί υπάρχουν θέματα που δεν έχουν επιληθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ευρύτερη προσέγγιση προς το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν και καλούμε και το Καρτούμ και την Τζούμπα να αναζητήσουν τη Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κυρίως στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, της δημιουργίας δυνατοτήτων, της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών και της θέσης των γυναικών. Ε, προσπαθούμε από κοινού με τα κράτη-μέλη να προσφέρουμε ε, την βοήθειά μας ε, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στόχο έχουμε να συντάξουμε μια έκθεση δίνοντας σημασία στην παιδεία, στη διαχείριση δάτων στη δικαιοσύνη, στο κράτο δικαίου, ε, στην αστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση του Νοτιού Σιντάν για να εφαρμοστεί έγκαιρα το συμφωνή, η Συμφωνία Κοτονού ω πλαίσιο τη βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ είμαι σε στενή επαφή με τον Νότιο Σουδάν ε, τόσο στι Βρυξέλλες όσο και στη Τζούμπα. Ελπίζουμε ότι τα μέλη τη Συμφωνία Κοτονού θα βοηθήσουν και αυτά ώστε να υπάρχει διαθρωμένος διάλογο με τη νέα κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν. Εν τω μεταξύ Ένωση θα συνεργαστεί στενά με τα Ηνωμένα Έθνη για να υποστηρίξει την κυβέρνηση του Νοτιού Σιντάν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πρόγραμμα δημιουργίου κράτου ε, και επίτευξη ειρήνη, ε, κυρίω μετά την εντολή των Ηνωμένων Εθνών. Να υπάρξει μια μεταβατική κατάσταση, μια συμφωνία με την κυβέρνηση του Νοτιού Σιντάν. Όλοι μα προσβλέπουμε στο να συμμετάσχουμε σε μια μεγάλη διεθνή διάσκεψη για τον Νότιο Σιντάν που θα λάβει χώρα κατά τα τέλη του έτου στην Ουάσιγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να έχει επιτόπου εκπροσώπους έτσι ώστε να είμαστε αξιόπιστοι. Επιθυμούμε το γραφείο μας στην Τζούμπα να το μετατρέψουμε σε κανονικό γραφείο εκπροσώπησής μας ε, το στομό των δυνατών, να έχουμε επιτόπου τις απαραίτητες δυνατότητες για να μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εξάλλου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών αναπτύσσοντας ε, συνδέσμους με την ε, νομοθετική συνέλευση του Νοτιού Σιντάν. Ενώ εστιάζουμε την προσοχή μας στο Νότιο Σουδάν, δράτω με τις ευκαιρίες για να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση στο Βορρά, στο Σουδάν και αυτή μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Συνεχίζεται η σύραξη ανάμεσα στις ε, αντιμαχόμενες ε, φυλές ε, πάνω από 300.000 άνθρωποι αναφέρεται ότι έχουν εκτοπιστεί και μέχρι τώρα δεν επιτρέπεται στις ανθρωπιστικές οργανώσεις η πρόσβαση. Ελπίζω ότι θα βρεθεί χώρος για να, χρόνο για να συντηθεί και η κατάσταση στο Σουδάν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Τυρολιάν, θέλετε να καταλήξετε. Α, όχι, συγγνώμη, την κυρία Ντεκάιζερ ξέχασα, την κυρία Ντεκεζέρ μάλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ουσιαστικά τα ερωτήματα που έχω Απευθύνω την κυρία Μάρστιν, η οποία νομίζω ότι έχει πιο πρόσφατες πληροφορίες. Η έκθεση την οποία μας ανέφερε ο Πατρίς ε, Τυρολιά, νομίζω ότι είναι ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο ε, μιας συγκεκριμένης ε, χρονικής στιγμής. Αλλά η κατάσταση εξελίσσεται. Υπάρχει αυτή η νέα δημοκρατία που γεννήθηκε, πρέπει να τη στηρίξουμε όπως λέει η κυρία Μάρστεν. Σίγουρα έγινε ε, το πρώτο βήμα με την ανεξαρτησία και ό,τι έχει αποκολουθήσει, αλλά πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμη βήματα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το γεγονός ότι θα έχουμε ένα στρατηγικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρονται κάποια ζητήματα που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και σε ποιο πλαίσιο μπορούμε να βοηθήσουμε τον Νότιο Σουδάν να αναπτυχθεί. Και φυσικά είναι και πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τον Νότιο Σουδάν στον στρατηγικό σχεδιασμό. Ουδόλου σε εύκολο εγχείρημα. Έχω κάποιες παρατηρήσεις ε, προς το παρόν τουλάχιστον. Πρώτη παρατήρηση, ερώτηση που βρίσκεται, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η φάση ανάπτυξης ε, του συντάγματος, πώς προχωρεί το νομοθετικό έργο που είχε δημιουργήσει και κάποιες μικροεντάσεις μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος ε, και του κόμματος της αντιπολίτευσης ε, στο Νότιο Σουδάν. Η αντιπολίτευση γνωρίζουμε ότι είχε αυτό, αυτό... συγγνώμη από το νομοθετικό αυτό έργο. Πότε πιστεύετε ότι επίση θα γίνουν εκλογές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο εκρεμούσε τον Ιούλιο. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να ξέρουμε αν έχουμε κάποιες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Δεύτερο ερώτημα. Ναι, πράγματι, αυτά που είπατε για τη Συμφωνία του Κοτών είναι πολύ σωστά. Το Νότιο Σουδάν είναι έτοιμο να επικυρώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού. Ξέρουμε τι γίνεται με τον Βόρειο Σουδάν, με τον Μπασίρ. Ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Συμφωνία επίσημη δεν υπήρχε, αλλά μεταξύ Σαλμπακύρ και Μπασίρ υπήρξε μια συμφωνία κυρίων πριν τον Ιούλιο. και μάλιστα είχε πει ότι θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής ε, του Μπασίρ ε, ε, γιατί θέλω να κρατήσω καλές σχέσεις με τον Βορρά. Ο πιο λοιπόν μεγάλος υποστηρικτής του στο θέμα του ποινικού δικαστηρίου είχε πει ο Σαλμπακή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το θέμα και θα ήθελα να επιληφθεί όχι μόνο η δική μα Επιτροπή, ίσω και η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα μπορούσαμε ίσω να έχουμε μια συζήτηση στο πλαίσιο των κατεπηγόντων για την κατάσταση ε, στα όρη Νούμα, Νούμα Mountains. Η Ρόζαλντ Μάρστεν μας είπε ότι υπάρχουν 300.000 εκτοπιστέντες, βομβαρδισμοί, ε, πρόβλημα με τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, καταστροφική κατάσταση. Και σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για το βόρειο Σουδάν δεν έχουμε ολοκληρώσει το Comprehensive Peace Agreement, γιατί δεν υπήρξαν διαβουλεύσεις ε, μεταξύ το Blue Nile και το South Cordovan. Και ξέρουμε ότι ελοχεύουν κίνδυνοι για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κατεπήγον από πλευράς ανθρωπιστικής ισχύει, τι πιέσεις όμως μπορούμε να ασκήσουμε στο βορρά, στο βόρειο Σουδάν. Γιατί δεν ξέρω αν έχουμε πολλούς μοχλούς άσκησης πίεσης, θα μας πείτε εσείς τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε στο νότο, μπορούμε, στο βορρά, συγγνώμη, μπορούμε να πιέσουμε τον Μπασίρ να σταματήσει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και σε ό,τι αφορά τον Νότο, τον Νότιο Σουδάν να βοηθήσουμε την πορεία του προς τη δημοκρατία και να μην περιμένουμε τις προσεχείς εκλογές. η κατάρτιση και όλα αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η πρόεδρος, ωραία, λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο, στον κύριο Γκαρίδο Λουίς από την Κομισιόν, εφόσον επιθυμεί να μιλήσει. Αν όχι, να δώσω τότε το λόγο στην κυρία Μάρστεν. Γιατί νομίζω τα ερωτήματα απευθύνονταν σε εσά πιο πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση ε, σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει τώρα ε, ως προς το Σύνταγμα, υπήρξε μια διαδικασία Προετοιμασίες και σύνταξης ε, ενός ε, προσωρινού συντάγματος, το οποίο, όπως ε, πολύ σωστά είπατε, έδωσε τη προκάλεσε ένταση με την αντιπολίτευση, η οποία αντιπολίτευση ε, θέλησε στη διαδικασία αυτή να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό λοιπόν το προσωρινό σύνταγμα εγκρίθηκε πριν από τις 9 Ιουλίου και οι επόμενες φάσεις ε, για την προετοιμασία μόνιμου συντάγματος με τον Νότιο Συντάν έχουν ήδη ξεκινήσει και εμεί ε, ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση του Νοτιού Συντάν να διασφαλίσει ότι σε αυτή την επόμενη φάση θα υπάρξει μια ευρεία διαδικασία αναθεώρησης του προσωρινού συντάγματος στην οποία ε, θα συμπεριληφθούν ε, τα κόμματα της αντιπαλίτευσης η κοινωνία των πολιτών και πολλοί άλλοι. Όσον αφορά τώρα τη Συμφωνία Κοτονού, είμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν για να διασφαλίσουμε ότι η κυβέρνηση εφόσον ε, το επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία, πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Το, η γλώσσα στη Συμφωνία Κοτονού, το θέμα ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αυτά η κυβέρνηση της Τζούμπα πρέπει να τα λάβει υπόψη της και είναι σημαντικό να δουν και τα υπέρ και τα κατά του όλου θέματος. Πάντως, αν τελικά αποφασίσουν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν ε, με τη Συμφωνία Κοτονού, αυτό μοιάζει να διαφαίνεται, είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για να τους βοηθήσουμε ε, να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στον κύριο Τυρολιά, ο λόγος τον κύριο Ρινάλνη, ο οποίος ζήτησε να μιλήσει. Κυρία Πρόεδρε, συμπληρώνω την ενημέρωση του κυρίου Τριολιάν, τον οποίο ευχαριστώ, που προείδρευσε τις αντιπροσωπίες μας. Λυπάμαι, δεν ήμουν εδώ όταν έλαβε το λόγο, αλλά έπρεπε να είμαι σε παράλληλη συνεδρία, είχαμε ψηφορίες καθώς και συντονιστές. Λοιπόν, θέλω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, ο ρόλος των ΜΚΟ. Το Νότιο Σουδάν είναι μια χώρα που το κράτος είναι αδύναμο. Οι έχουν ισχυρή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή. Σήμερα ο ρόλος τους πρέπει να γίνει αντικείμενο αναθεώρησης, διότι έχουν πλέον να τα βάλουν πέρα με ένα κράτος. Υπάρχουν συνθήκες δηλαδή που δεν συνέτρεχαν στο παρελθόν. Πρόκειται για πρόκληση για τη ΣΜΚΙΟ. Αφιερώσαμε σχεδόν ένα ολόκληρο απόγευμα πάνω σε αυτό το θέμα με τη ΣΜΚΙΟ. Πρέπει δηλαδή να προσαρμοστούν σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και το νέο κράτος όμως, του νέου Σουδάν, πρέπει να αξιοποιήσει το ρόλο, την γνώση και την εμπειρία στην πράξη επιτόπου αυτών των ΜΚΟ στην διαβίβαση της ε, βοήθειας και στην παροχή βασικών υπηρεσιών. Δεύτερον, έχουμε εννοείται το πρόβλημα με τον Βορρά, αλλά έχουμε και το πρόβλημα το εσωτερικό, της εθνικής συμφιλίωσης, που είναι πρόβλημα προτεραιότητας. Γιατί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο Βορρά υπάρχουν αντιπαλότητες ε, εξαιρετικά οξυμένες ακόμη και σήμερα, οι οποίες απαιτούν συμφιλίωση για να δημιουργηθεί μια συναντήληψη περί συνύπαρξης, ελληνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Αυτό, επαναλαμβάνω, αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την κυβέρνηση τη Τσούμπα όσο και για την διεθνή κοινότητα. Τρίτον, εξίσου σημαντικό, ο κύριος Πόρος στον Αντισουδάν είναι το πετρέλαιο, αυτό το γνωρίζουμε επιμείναμε στην αξιοποίηση της εμπειρία του Ανατολικού Τιμόρου, που δημιουργήθηκε ένα ταμείο στο οποίο κατατίθενται τα έσοδα από τις πωλήσει πετρελαίου. Είναι ένα ανεξάρτητο από τον κρατικό προπολογισμό και αυτό ακριβώ εξασφαλίζει διαφάνεια στη χρήση των σχετικών πόρων. Αυτό πρέπει να αποτελέσει και μια προϋπόθεση για την πρόληψη κάθε είδους διαφθοράς. Μίλησαμε και με βουλευτές οι οποίοι είναι ταγμένοι στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Από τη στιγμή όμως που θα φτάσουν στα χέρια τους τα πραγματικά έσοδα από το πετρέλαιο, ε, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε λόγο όλα αυτά, είχαμε και προτάσεις και καλές πρακτικές να γιατί όπως είπε το Ανατολικό Τιμόρ είναι ένα αξιόλογο προηγούμενο. Γι' αυτό και επιμείναμε ε, να γίνει κάτι αντίστοιχο ε, στις αρχές της Τζούμπα. Κύριε αν θέλετε τον λόγο μήπως ξανά. Παρακαλώ, χωρίς μικρόφωνο. Απλώς... Πολύ απλά για να ολοκληρώσω, πιστεύω ότι η χώρα αυτή είναι μια χώρα η οποία προκαλεί πολύ ενδιαφέρον και πολλοί θέλουν να, να βοηθήσουν ώστε να κερδιθεί το στίχημα της ανάπτυξης. Έχει πολλούς ε, φυσικούς ε, πόρους, ε, ορυκτό πλούτο, ύδατα στο Νότιο Σουδάν, αλλά δυστυχώς υπάρχουν εντάσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Υπάρχει εκμετάλλευση από το Βόρειο Σουδάν, κάτι που αυτή την τελευταία πενικονταετία ε, απογύμνωσε ε, τη χώρα, την απομίζησε. Επομένως έχουμε ακόμα πάρα πολλές προκλήσεις ε, να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορώ να δεχθώ τη διαπίστωση που γίνεται σήμερα ότι δεν θα επιτευχθούν ποτέ οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Είναι μια διαπίστωση που, στην οποία προέβη ο ΙΕ λέει ότι τι τις παρούσες συνθήκες δεν θα επιτευχθούν ποτέ οι αναπτυξιακοί στόχοι της ε, χιλιετίας. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί ώστε το Νότιο Σουδάν να είναι ένα παράδειγμα επιτυχίας και όχι αποτυχίας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τυρολιά. Μπορούμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Πολιτική γειτονία. ανταλλαγή απόψεων ε, για μια δική μου γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια επί της ουσίας για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και αν μου επιτρέψετε θα μου δώσω το λόγο για να σας παρουσιάσω εν συντομία το σχέδιο γνωμοδότησης. Λοιπόν, το σχέδιο έκθεσης της ΑΦΡ για την αναθεώρηση ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας ε, είναι άρτιο, είναι ισορροπημένο και το προσυπογράφω ως προς το περιεχόμενό του. Απλά θα ήθελα να λάβει υπόψη η Επιτροπή κάποιες σκέψεις που είναι σημαντικές ε, για εμάς στην Επιτροπή Ανάπτυξης και δεν υπάρχουν ακόμη αυτά τα στοιχεία. Και ε, θα προσπαθήσω να τα αναφέρω αυτά τα σημεία στο σχέδιο γνωμοδότησης, όπου επιμένω σε κάποια σημαντικά σημεία όπως είναι η συνεκτικότητα πολιτικών υπέρ της ανάπτυξης, κάτι το οποίο πρέπει να φαίνεται γιατί είναι και μια σημαντική ε, ανησυχία της Επιτροπής μας. Πρόκειται άλλωστε για συνταγματική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίζεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και στις, ε, στην Ανατολική και στην νότια εταιρική σχέση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη λοιπόν αυτή την υποχρέωση. Έτσι στην γνωμοδότησή μου λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους ε, της αναπτυξιακής συνεργασία κατά την υλοποίηση τη πολιτική γειτονία και ειδικότερα τον βασικό στόχο που είναι η μείωση και διεκρίζωση της στόχιας. Επίσης θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αναφέρεται στην γνωμοδότησή μου το θέμα των μεταναστευτικών ροών ή σχέσεων ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονικών χωρών από την νότια και ανατολική εταιρική σχέση και δεν θα πρέπει τις σχέσεις αυτές να τις βλέπουμε μόνο υπό το πρίσμα ε, των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας. Αυτές οι μεταναστευτικές σχέσεις πρέπει να αναλυθούν και στο πλαίσιο της βιώσιμη σταθερή ανάπτυξης ε, των γειτονικών μας χωρών. Έτσι, στη γνωμοδότησή μου καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΑΣΕ να επικεντρώσουν τι μελλοντικέ του πολιτικές στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων και όχι μόνο στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Εκτιμώ επίσης ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο προπολογισμό τη αναπτυξιακή βοήθεια και τη ανθρωπιστική βοήθεια σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναδιατίθενται για τη χρηματοδότηση τη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Μιλώ επίση για την λύπη την οποία εκφράζει η Επιτροπή μα σε σχέση με την κατάσταση στην Αγγή Ανατολή, βλέποντα ε, την ανθρωπιστική κατάσταση και την ανθρωπιστική βοήθεια, την πολύ σημαντική που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ ε, την περιοχή αυτή και κυρίω προ την ε, Ούνρα. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΑΣΕ να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ένα πολιτικό και διπλωματικό εταίρο πρώτη κατηγορία στην Αγγή Ανατολή και ολοκληρώνοντα, υπενθυμίζω ότι η Αραβική Άνοιξη έχει σημαντικέ επιπτώσει στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τι γειτονικέ τη χώρε. Θέλω να επιμείνω λοιπόν ε, στη στήριξη προ την τοπική κοινωνία των πολιτών που κατάφερε να χειραφετηθεί, να απεξαρτηθεί από την εξουσία εκεί. Η χειραφέτηση αυτή όμω θα πρέπει να συνοδευτεί με πραγματική δημοκρατική πρόοδο και ε, με το μεγαλύτερο σεβασμό των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ειδικά δικαιώματα των γυναικών, σεβασμό στη δικαιοσύνη και του κράτους δικαίου, θεμελιώδεις ελευθερίες και χρηστή διακυβέρνηση, η δίκαια κατανομή των ε, εσόδων και εισοδημάτων και καταπολέμηση της φτώχειας ε, που πλήττει αυτά τα κράτη. Σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας. Ο κύριος Γκερέρο είναι ο πρώτος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η καλύτερα κυρία Προεδρεύουσα, μόνιμα εισηγήτρια για την ανθρωπιστική βοήθεια, ε, συντάκτρια γνωμοδότησης για τη συγκεκριμένη έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Διάβασα με προσοχή τη γνωμοδότησή σας και συμμερίζομαι τις ε, απόψεις και τα σημεία τα οποία αναφέρεται και σε ό,τι αφορά την διασύνδεση της αναπτυξιακής πολιτικής με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά και σε ό,τι αφορά τη διατήρηση για την ανάπτυξη των πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη. Δηλαδή να μην υπάρχει σύγχυση με κονδύλια της πολιτικής γειτονίας. Συμφωνώ επίσης με αυτό που είπατε ότι είναι ανάγκη να έχουμε έναν ενεργητικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, Εγγύης Ανατολή και να έχουμε μια κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό και πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία στα προβλήματα σε αυτή την ε, γεωγραφική περιοχή. Θέλω να επισημάνω ότι Μεταξύ των φαινομένων που βλέπουμε στον κόσμο να διαδραματίζονται τελευταία χρόνια, ίσως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα είναι η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, διότι μέσα σε τόσες καταστροφές, στην οικονομική κρίση, εν μέσω κοινωνικών επιπτώσεων πολύ αρνητικών σε ολόκληρο τον κόσμο, βλέπουμε ότι αρκετές χώρες ε, κοινωνίες ε, ιστορικά και παραδοσιακά καταπιεσμένες ε, ε, ακολούθησαν πλέον το δρόμο της δημοκρατικής μετάβασης και της ελευθερίας. Δεν έχει ολοκληρωθεί η πορεία, είμαστε ακόμη σε πλήρη εξέλιξη της όλης διαδικασίας, εξού και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη δέσμευση να βοηθήσει, να συνοδεύσει αν θέλετε τις χώρες αυτές στην πορεία τους, στη δημοκρατική και πολιτική μετάβαση. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική και η Νότια Μεσόγειος, η νότια εταιρική σχέση. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πάντοτε πόσο σημαντική είναι αυτή η περιοχή και η νότια εταιρική σχέση, γιατί μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τον ενεργειακό εφοδιασμό, την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια. Και η σημασία της περιοχής υπήρχε και από πριν, αλλά τώρα είναι ακόμη πιο σημαντική γιατί ε, θα βρίσκεται στο μέσο αυτών των δημοκρατικών ε, δομών που δημιουργούνται. Εμεί πρέπει να βοηθήσουμε στη δημιουργία των δημοκρατικών δομών και πρέπει να βοηθήσουμε και μέσω τη αναπτυξιακή πολιτική. Επομένω, η συνολική εστίαση τη έκθεση, δηλαδή ότι η αναπτυξιακή πολιτική την οποία προσπίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, το να γίνει λοιπόν αυτή η πολιτική ένα απαραίτητο εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό επιχείρημα. Θα ήθελα επίσης να λάβετε υπόψη σας, αν μπορείτε να το προσθέσετε, κάτι το οποίο είναι συχνό στην Επιτροπή μας, δηλαδή σχέση, διασύνδεση της φάσης αποκατάστασης, ανοικοδόμησης, ιδίως στις χώρες εκείνες όπως τη Λιβύη για παράδειγμα, όπου υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση και οδηγεί σε σημαντικές καταστροφές, όχι μόνο στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά και στις ε, καταστροφές ε, των υποδομών. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε επιπλέον αναφορά στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για την Νότια Μεσόγειο που θα παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες πολιτικής μετάβασης κατά κάποιο τρόπο ζητούμε να συμπεριληφθεί στη δράση του ειδικού αυτού απεσταλμένου ο τομέας της ανάπτυξης. Ο κύριος Μπερναρντίνο Λεόν είναι ο ειδικός απεσταλμένος. Και φαντάζομαι ότι θα είναι απόλυτα διατεθειμένος ε, να αναλάβει και έναν ρόλο ε, προώθησης ε, της αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό το οποίο βλέπουμε να συνοδεύει τη μετάβαση ε, των χωρών αυτών είναι η κινητοποίηση των νέων και των γυναικών και η επιθυμία για ελεύθερες εκλογές. Νομίζω ότι ένα μέρος της αναπτυξιακής μας πολιτικής θα είναι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών, γυναίκες, νέοι, και βέβαια θα πρέπει να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε και τα κοινοβούλια. Όταν ε, προκύψουν βέβαια, γιατί μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε εκλογές σε χώρες που έχουν μικρή ε, κοινοβουλευτική εμπειρία και ε, εμπειρία από εκλογέ. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τις διαδικασίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεοχάρου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, αυτά που έχετε γράψει στη γνωμοδότηση με εκφράζουν απόλυτα και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την αρτιότητα. Θέλω να προσθέσω ένα σημείο όσον αφορά την διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχετε πει ότι δεν πρέπει να μας νοιάζει μόνο η διαχείριση της κρίσης όποτε εκδηλώνεται αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων στην συνέχεια. Ωστόσο, εδώ θέλω να επισημάνω ότι εφόσον μιλάμε κατά μείζωνα λόγο και για τις χώρες που δέχονται το κύριο κύμα των προσφύγων θα πρέπει να γίνεται ένας επιμερισμός ανάμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του του οικονομικού φορτίου για την προστασία των προσφύγων και των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι δυνατόν τα φτωχά κράτη του Νότου που δέχονται και τη μεγαλύτερη πίεση να αντέχουν όλο αυτό το ε, οικονομικό φορτίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, κ. Τρεμονίνη. Thank you very much. Yes. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι... Um, ε, νομίζω ότι η έκθεση επισημαίνει τα βασικότερα θέματα και θα ήθελα απλά να σας υπενθυμίσω ότι οι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας είναι η σταθερότητα, η ευημερία, ε, επί τη βάση ή για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους και οι κοινοί στόχοι αφορούν την πραγματική δημοκρατία. Τα γεγονότα λοιπόν στην ε, Αραβική Άνοιξη κατέδειξαν ότι την σταθερότητα και την ευημερία μπορούμε να την επιτύχουμε μόνο εφόσον υπάρχει ε, δημοκρατία και αυτό νομίζω το γνωρίζουν όλοι. Τώρα, θα ήθελα να πω επίσης ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας έχει ως στόχο να ε, προάγει την σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία, δημιουργώντας το πλαίσιο, θα λέγαμε, και βοηθώντας ε, την κοινωνία των πολιτών να υπάρξουν θεσμοί που είναι απαραίτητο για να λειτουργεί η δημοκρατία. Να υπάρχει και κράτος δικαίου που είναι προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν η ευημερία έχει άμεση σχέση όπως ξέρετε με την παραγωγή προϊόντων. Οι στόχοι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με τους ε, στόχους της ε, ανάπτυξης. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτές τις ε, δύο πολιτικές. Ε, όσον αφορά τώρα στη μετανάστευση, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε και να προάγουμε τη σχέση ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Ε, τα μέλη μας ε, λοιπόν γνωρίζουν ε, πολύ καλά ότι διαπραγματευόμεθα τις συνεργασίες κινητικότητας και δυνατότητας μετακίνησης. Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις ε, στη Νότια Μεσόγειο, με την Τινησία και το Μαρόκο για να συσταθούν ε, συνεργασίες οι οποίες θα εξετάσουν και τους τρεις βασικούς πυλώνες της μετανάστευσης συμπεριλαμβανομένης και τις σχέσεις ανάμεσα στην μετανάστευση και την ανάπτυξη. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εμβάσματα ε, για την ανάπτυξη της χώρας προέλευσης, παραδείγματος και εμείς αυτό το κάνουμε, το προάγουμε. Αναφέρθηκε επίσης ότι θα πρέπει να ξεστούν θέματα ανάπτυξης και από την πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία θα πρέπει πάντα να έχει στόχους, ε, τους στόχους της ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή πολιτική ε, κατ' ουσίαν έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη των γειτόνων μας. Το μόνο το οποίο ίσως μπορούμε να συζητήσουμε είναι πώ ακριβώ θα επιμεριστούν τα αναπτυξιακά κονδύλια στα διάφορα μέρη του κόσμου. Βεβαίω και αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης, αλλά η πολιτική γειτονία σαφώς και έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη των γειτόνων μας. Ο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Μόλτ. Όχι, ναι. Ευχαριστώ για την κοινωνία των πολιτών. Να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη κάνει πολλά στην περιοχή. Υπάρχει ένα σχετικό μηχανισμό υποστήριξης που καλύπτει την Ανατολική και τον Νότο με στόχο την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την υποστήριξη τη δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί μηχανισμοί υποστήριξης της ανάπτυξης στην περιοχή. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τα συμπεράσματα αυτά. Να υπενθυμίσω ότι προθεσμία πολλής τροπολογιών είναι 14 Οκτωβρίου στις 12, 14 Οκτωβρίου στις 12. Η συζήτηση θα λάβει χώρα στις 7 Νοεμβρίου. Περιμένω σχόλια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να προσθέσετε. Δημοσιονομικός έλεγχος της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ που διαχειρίζεται η ΕΚΟ. συναδελφοί, για το θέμα αυτό. Στις 8 Δεκεμβρίου θα εγκριθεί το σχετική, η σχετική απόφαση. Μισό λεπτό γιατί τα έχω μπλέξει λίγο, λέει ο Πρόεδρος. Ως εισηγητριά γνωμοδότησης, δίνω το λόγο στον εαυτό μου για μια σύντομη παρουσίαση της, του σχεδίου γνωμοδότησης. Έχω δύο διαφορετικούς ρόλους σήμερα η αρμόδια επιτροπή δεν θέλησε να δώσει το σχέδιο γνωμοδότηση, αλλά η γραμματεία μα ενημέρωσε για κύρια στοιχεία τουλάχιστον, τα οποία έχουν ω εξή. Η ανάλυση τη Επιτροπή Ελέγχου των Προπολισμών σχετικά με το σύστημα χρηματοοικονομικού ελέγχου έχει καταληξεί σε θετικά συμπεράσματα κάποιες επικρίσεις υπήρχαν για το 2009 όσον αφορά το σύστημα αναφοράς και ιστορικού ελέγχου των ε, οργάνων των ΕΕ που είναι τέρη της Γενικής Διευθύνσης ΕΚΟ όσον αφορά τη συνεργασία με τη ΜΚΟ ο κ. Μαρτά μας λέει ότι χρειάζονται βελτιώσεις όσον αφορά την σύναψη συμβάσεων και την διαχείριση κινδύνου, την διαφάνεια όσον αφορά τους υπεργολάβους, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο η Γενική Διεύθυνση χειρίζεται τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τον προπολογισμό για τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερος ρεαλισμός στην εκτίμηση των δαπανών και ότι ο προπολογισμό αυτός πρέπει να ενισχυθεί. Τέλος, όσον αφορά τις πρόσφατες κρίσεις στην Αϊτή και στο Πακιστάν, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή τη για την ταχύτατη και ουσιαστική απάντηση τη γενική διεύθυνση ακόμη και σε πολύ δύσκολε συνθήκες. Εκφράζει όμω τη λύπη τη για την ε, αδυναμία της παρεμβασή μα, Υπογραμμίζει την έλλειψη επαρκούς προπολογισμού για τις ανθρωπιστικές παρεμβάσει. Αυτό στο παρελθόν δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα εξέβρεση πόρων, κυρίω προ το τέλο τη χρονιά, όταν τα σχετικά κονδύλια έχουν εξαντληθεί. Στην γνωμοδότηση εκφράζω επίση την ικανοποίησή μου για την αύξηση των κονδυλίων για την ανθρωπιστική βοήθεια και για το αποθεματικό έκτακτη βοήθεια που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2004-2020 έως και 813 εκατομμύρια εκατομμύρια σε σύγκριση με την ε, περίοδο 7-13. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και απρόβλεπτες κρίσεις. Επίσης ε, έγινε πρόοδος την εκτακτή βοήθεια, στην αποκατάσταση ζημιών και την ανάπτυξη. Είμαστε πλέον πιο ευέλικτοι σε σχέση με τους παλιότερους δημοσιονομικούς κανόνες. Επίσης, στην πτώση κρίσης, η μεταφορά κονδυλίων από τη μία θέση στην άλλη, παρά το ότι προβλέπεται εν γέννη, παραμένει δύσκολη. Χαίρομαι γιατί το 2012 θα οργανώσουμε και μία σχετική ακρόαση. Επίσης, σχολιάζουμε τα εργαλεία της Γενικής Διεύθυνσης και την επιλογή των έργων είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή υποψηφίων έργων Έχουμε μια καινοτομία λοιπόν μπροστά μα, η οποία θα κάνει τη δράση μας πιο αποτελεσματική και ταχύτερη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να φροντίσουμε αυτή η καινοτομία να μην αποκλείσει μικρέ ΜΚΟ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που πολλές φορές ε, έχουν περιορισμένες διοικητικές δυνατότητες. Τάσουμε επίση υπέρ τη ε, διατήρηση ποικιλία συνεταίρων και συνεργατών, ιδιαίτερα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Γενική Διεύθυνση επιλέγει πολύ προσεκτικά τους εργάτες τη, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα βάσει πρακτικών και κανόνων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ποιότητα των εταίρων είναι αναμφισβήτητη, γίνεται τακτική έλεγχη των πόρων μέσω ιδιωτικών ελεγχτικών εταιριών οι οποίες ε, θεμητοποιούν και την δράση μας στον ανθρωπιστικό τομέα ο λόγο σε εσά, αλλά δεν βλέπω κάποιον να θέλει τον λόγο. Κυρία Κέλλερ. Μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι σχετική. Όμως... Ε, ο έλεγχος του προϋπολογισμού ε, λέει ότι στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, καταποκοπή ποσά, εφάπαξ ποσά, γιατί αλλιώς ε, είναι δυνατόν να υπάρξουν και πάρα πολλά λάθη. Τώρα τι έγινε αυτό, αυτό το αφαιρέσατε από την έκθεση ή μήπως δεν είναι σημαντικό για τον τομέα της υπηρεσίας ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ακριβώς έγινε. Καλό ερώτημα. Τι πιστεύετε κύριε Γκέρνης εσείς. Je Να δώσω το λόγο στον κύριο Σπίγκελε από την ΕΚΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να αντιδράσω έτσι σύντομα όσον αφορά το σχέδιο της έκθεσης. Εμείς τη χαιρετίζουμε, τη θεωρούμε σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα ισόρροπη. Αναγνωρίζουμε απόλυτη σαφήνεια την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζει τα συστήματα ελέγχου, αυτό το να έρχεται αυτό σαν αναγνώριση από την Επιτροπή Προλογισμών είναι ιδιαίτερο κοπλιμέντο για μας ε, όπως αναφέρατε, υπάρχουν αρκετά θέματα, αναφέρονται αρκετά θέματα, τα οποία βέβαια χρήζουν ε, περαιτέρω εξέτασης. Κυρίως ε, όσον αφορά ε, την κατάθεση εκθέσεων και την επαλήθευση των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Η εξέταση συνεχίζεται, αλλά πρέπει να υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας. Και τέλος, η έκθεση αναφέρεται στο θέμα του δημοσ... της ενίσχυσης του προϋπολογισμού. Η έκθεση που έχω μπροστά μου δεν ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα την ΕΚΟ. Υπάρχουν κάποιες ε, δαπάνες όπου ίσως θα μπορούσαμε πράγματι να έχουμε καλύτερα ε, καταποκοπή ποσά. Αλλά όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, εμείς δουλεύουμε πάνω στις πραγματικές δαπάνες. Άρα δηλαδή αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι θέμα προτεραιότητας. Ε, και όσον αφορά στις ε, συστάσεις, εδώ έχουμε μπροστά μας δύο σημαντικές εκθέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κουραστήκατε, βλέπω, δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμή κατάθεσης ε, των τροπολογιών έχει τροποποιηθεί. 12 Οκτωβρίου πλέον, λίγη στις 5 το απόγευμα. Και η ψηφοφορία θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο 19, τα διάφορα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Επομένως, η ημερομηνία της προσεχικούς συνεδρίασής μας στις Βρυξέλλες 7 Νοεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Η συνεδρίασή μας θα συνεχιστεί το απόγευμα σήμερα με τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση των Επιτροπών Ντέβη και Ντρουά με τα Εθνικά Κοινοβούλια θέμα θα είναι η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αναπτυξιακή πολιτική. Σας προσκαλώ όλες και όλους να συμμετάσχετε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρούσες όταν έρχονται συνάδελφοί μας, ομόλογοι μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια για να συναντηθούν με εμά εδώ. Καλή όρεξη λοιπόν και θα τα πούμε το μεσημέρι. Κύριε Μπέρμαν, τώρα που ήρθατε, Vous revenez à 15h, monsieur Berman. Να ελάτε στις 3 με τους εθνικούς βουλευτές.